αποφάσισαν να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις βάσει του άρθρου 69C, παράγραφος 1 του κανονισμού. Οι εκθέσεις ε, που αποτελούν και εντολή για τις ε, διαπραγματεύσεις αυτές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ε, Σολομέλειας και οι τίτλοι του θα δημοσιευθούν στα πρακτικά της παρουσιά.